υποβάλουμε προτάσεις στο, στο άμεσο μέλλον ε, για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε αυτές τις παράνομες μεταφορές οξυγόνων προβλήτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ όσους έμειναν μέχρι τα μεσάνυχτα. Α, ξέρετε υπάρχει αυτή κάπως χαλαρή πειθαρχία στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται αύριο 11 Μαΐου από τις 9 το πρωί. Η ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Εύχομαι συναδέλφους καλή